αλλόμενα μέρη δηλαδή. Είμαι πεπισμένος ότι έτσι θα βοηθήσουμε αρκούντος τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε Μπαρνιέ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση σε αυτό το σημείο. Το επόμενο σημείο είναι οι παρεμβάσει σε ενός λεπτού σύμφωνα με το, με το άρθρο 150 του κανονισμού. Ε, ο κύριος Κούκαν έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτά τα έγγραφα τα οποία πρόσφατα έχουν δημοσιευθεί από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν την διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δώσει το μήνυμα στι χώρε που θέλουν να υποβάλουν την αίτηση ένταξη για το ότι η πρόοδο γίνεται μόνο επί τη βάση πραγματικών επιτευγμάτων, πραγματικών επιδόσεων. Οπότε, σύμφωνα με όλα αυτά, εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τι μεταρρυθμίσει ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι διαπίστωσαν ότι πάρα πολύ συχνά ακόμα και μετά από πάρα πολύ σημαντικού συμβασμούς είχαν πετύχει πάρα πολύ σημαντικά και οι υπόλοιποι απλώς έκαναν επίδειξη δύναμης αντί για κάποιο δημιουργικό διάλογο. Οπότε ε, τελικά ήταν θέμα χρόνου. Επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντική η πληροφορία το ότι θα πρέπει ε, τη δουλειά να την κάνουν οι ίδιες αυτές οι χώρες. Θα πρέπει, αν θέλουν να επιβάλλουν κάποια μέτρα στους πολίτες τους, θα πρέπει να επιδείξουν ε, κάποιες ε, επιδόξεις. δεν είναι δυνατόν κανείς να επικαλείται κάποιες μυστηριώδεις δυσκολίες. Δεν αρκεί αυτό. κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε. Σας ευχαριστώ Εάν πάμε για 30-40% ανεργία στους νέους σε ορισμένες χώρες και σε ορισμένες χώρες σχεδόν η μισή από τους νέους δεν έχουν δουλειά, τότε ε, κάτι θα πρέπει να γίνει σε εθνικό, σε κοινωνικό επίπεδο. Επίπεδο, ε, κατά τη δική μου γνώμη, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε πάνω σε προγράμματα απασχόληση. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα στα προβλήματα τη νεότητα. Θα πρέπει να βρούμε κάποια ε, μέτρα τα οποία να βοηθάνε το να βρουν δουλειά οι νέοι και θα πρέπει να παράσχουμε κάποιες κοινωνικές ε, εγγυήσεις ούτως ώστε τελικά να μπορούμε να δούμε ποιες είναι θέσεις εργασίας που ε, ε, προσφέρονται να δούμε πού χρειάζονται εργατικά χέρια όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ούτω ώστε να δούμε μέσα από την παιδεία, μέσα από κάποια προγράμματα δεξιοτήτων τι θα πρέπει να γίνει, επιχειρηματικό πνεύμα να καλύψουμε στους νέους τέτοιου είδους εκπαίδευση επιχειρηματική να ξεπηδήσουν νέες εταιρείες, να ενημερωθούν οι νέοι για το τι προγράμματα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιο είδους ε, στάζ, κάποιο είδους περίοδοι εκπαίδευσης. έχει λόγο. Αναγνωρίστηκε από την ΕΤΑ ότι απέτυχε η τρομοκρατία. Οπότε θα πρέπει να θυμηθούμε ότι οι Βάσκοι και οι Βάσκε ποτέ δεν θέλουν να, να αφαίρεται η ζωή από κάποιον. Το, το, 1978 έγινε το πρώτο συλλαλητήριο κατά τη ΕΤΑ, κατά τη τρομοκρατία ΕΤΑ. Και το, οι περισσότεροι στη χώρα των Βάσκων φώναξαν όχι στην ΕΤΑ. Τώρα έχουμε ε, την επικύρωση αυτού του προγράμματος για τη χώρα των Βάσων ξεκίνησε το 2010. Θα πρέπει μόνος έτσι να ενισχύσουμε την ειρήνη, να υπάρχει καλύτερη συμφιλίωση, συνύπαρξη, ούτως ώστε να μην επαναλάβουμε τα, τα κάποια λάθη του παρελθόντος. Οπότε θα πρέπει να σεβαστούμε το πόσο υπέφεραν τα θύματα, να ξεχάσουμε την εκδίκηση. Θέλουμε αλληλεγγύη, σεβασμό και δικαιοσύνη. Οπότε γι' αυτό σας λέω τώρα να κρατήσουμε κάποιο είδου ε, σιγή ή να του χειροκροτήσουμε εν πάση περιπτώσει αντί για τη ε, τα θύματα γιατί αξίζουν τη επικρότηση. Ευχαριστούμε κυρία Βιλμπάου Μπαράντικα. Ο κύριος Σουίνμπορν. Κυρία, συγγνώμη Σουίνμπορν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ε, συγχαρώ ε, για το, τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος στη Νέα Ζηλανδία ε, η ομάδα της Ουαλίας ε, πρέπει να αξίζει συγχαρητήρια για του, να, τις επιδόσεις τους ημιτελικούς. Ε, είναι πραγματικά ε, λόγος για να νιώθουμε μεγάλη περηφάνεια πραγματικά είναι παράδειγμα πώς οι αθλητές και οι αθλήτριες μπορεί να συμβάλλουν στην εθνική ενότητα και προαγωγή του πολιτισμού παγκοσμίω. Ο αθλητισμός είναι ε, πηγή περηφάνειας ε, στα ευρύτερα πολιτισμικά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιηθεί λοιπόν. Θέλω να συγχαρώ και πάλι ε, την ομάδα της Ουαλίας. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Σουίνμπερν. Και τώρα ο κύριος Σταβάρες. Ευχαριστώ. Τις τελευταίες εβδομάδες χάσαμε το 14% των ε, συντάξεων και συνολικά φτάσαμε σε μία απώλεια της τάξης του 30% των μισθών και των συντάξεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα χρέος που ανέρχεται στο 130% του ΑΕΠ και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές γίνονται δόλιες πτωχεύσεις από επιχειρήσεις για να μπορέσει κανείς να γλιτώσει τους φόρους και πολλές φορές είδαμε ότι οι επιχειρήσεις πήγανε από την Πορτογαλία, Πορτογαλία κήρυξαν πτώχευση και μετά μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε σε μια σωστή εναρμόνιση γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι, πρωτίστως γενναιόδοροι, χωρίς όμως να είμαστε άπλιστοι. Δυστυχώς είδαμε όμως ότι δεν ίσχυσε αυτό. Με τα πολεμικά και κανένας δεν κέρδισε από αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Τρενταφυλίδης έχει το λόγο. Πρόεδρε, η απελευθέρωση την περασμένη εβδομάδα του Ισραηλινού στρατιώτη Γκυλάς Σαλίτ από τη Χαμάς με αντάλλαγμα την αποφυλάκηση πέραν των χιλίων Παλαιστινίων κρατουμένων προκάλεσε και δικαίως αισθήματα χαράς και αισιοδοξία σε αφότερες τις πλευρές και όχι μόνο για να μετουσιωθεί όμως αυτή η αισιοδοξία σε θετικό παράγοντα χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις εκ μέρους κυρίως του δυνατού του ισραήλ που έχει τη δυνατότητα να προβεί σε συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. μπορεί να προχωρήσει στη σταδιακή άρση του αποκλεισμού της γάζας στη σταδιακή απελευθέρωση όλων των παλαιστινίων κρατουμένων στο πάγωμα των οικισμών και η χαμάς στον οριστικό τερματισμό της εκτόξευσης ρουκετών εναντίον του ισραήλ μόνο έτσι θα συμβάλει η προαναφερθής ανταλλαγή κρατουμένων στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την ελπίδα αυτέ να οδηγήσουν σε λύση. διαφορετικά η απελευθέρωση του σαλίτ με ανταλλαγή την αποφυλάκηση μεγάλου αριθμού παλαιστινίων κρατουμένων θα μπορούσε να ενθαρρύνει πράγμα που όλοι απευχόμαστε την απαγωγή και άλλων ισραηλινών στρατιωτών με την προσδοκία ανταλλαγή του με παλαιστίνιους που εξακολουθούν να κρατούνται στι φυλακέ. Ευχαριστώ κύριε Τριανταφυλλίδη. Ο κύριος Μοργάντη τώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, τις τελευταίες μέρες άκουσα να λένε πολλοί ότι η Κίνα θα είναι ο, σωτή, ο πιθανός σωτήρας του ευρώ και της Ευρώπης. Μυρολατρικός και ενθουσιώδης ο τόνος σε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Ρωτώ απλά, από πού και ως πού όμως η, Ευρώπη, η Κίνα πρέπει να βοηθήσει την Ευρώπη. Δεν θα ήταν αυτό σκοπός αυτή η βοήθεια. Δεν θα ήταν το τελευταίο θανάσιμο πλήγμα που θα μπορούσε να δώσει η Κίνα στη Δύση. Βλέπετε τι ωραία τα έχει σχεδιάσει η Κίνα. Ενώ η Ευρώπη τα έχει μεσάνυχτα για το πώς μπορεί να παρέμβει. Εγώ έρχομαι από το Πράτο που έχει το πιο υψηλό ποσοστό κινέζικου πληθυσμού στην Ευρώπη. Ήρθαν να μας βοηθήσουν. Ελέγχουν όμως σήμερα όλη την πόλη σχεδόν. Έχουν σχεδόν καταστρέψει την κοινωνία του Πράτο και την οικονομία της πόλης. Ευχαριστώ κύριε Μοργάντη. Για ένα λεπτό κυρία Τσιντεσλεύσκα. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά κράτη-μέλη, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ενέκριναν την Ευρωπαϊκή Κάρτα για τις πολυμελείς οικογένειες για να βοηθήσουν δηλαδή τις οικογένειες με πολλά παιδιά τους δίνουν διευκολύνσεις Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό ο οποίος να, να αναγνωρίζει το καθεστώς των πολυτέκνων οικογενειών. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να βραβεύονται οι πολύτεκνες οικογένειες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχα δηλαδή με αυτό που γίνεται σε εθνικό επίπεδο είναι θεμελιώδες να αναγνωρίζουμε την αξία των πολυτέχνων οικογενειών σε μια Ευρώπη η οποία γερνάει συνεχώς. Απευθύνω έκκληση στην Κομισιόν για να αρχίσει να δρά το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ κυρία Τσιλεύσκα. Επόμενος ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη διαθέτει τεράστιο βασικό πλούτο με ποικιλίε τις οποίες θα πρέπει να προστατεύσουμε. Όμως η αποψήλωση των δασών έχει πάρει καταστροφικές διαστάσεις. Στο Ρετεζάτε, στη Ρουμανία, είχαμε μία τεράστια αποψήλωση των δασών. Και αυτό οδηγεί σε υποβάθμιση του, της ποιότητας του εδάφους και εξαφάνιση χλωρίδας και πανίδας. Η Ευρώπη έχει ένα σύστημα για την εποπτεία των δασών, το οποίο όμως έχει τεράστια κενά. Χρειάζονται να αναλυθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δασών, βελτιώνοντας αυτή την νομοθεσία και να βελτιώσουμε και τις πρακτικές διαχείρισης και διοίκησης αυτών των περιοχών, τόσο ώστε όλοι να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον πλούτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούτας. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκάλαγκα, παρακαλώ συνάδελφε. Uh, τώρα με μικρόφωνο. Χτε έγινε η Σύνοδο Κορυφή και περιμένουμε τώρα την Τετάρτη. Μάλιστα, συναρπαστική στιγμή για την Ευρώπη και για το ευρώ. Θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι για ένα γενικό διακανονισμό για να επιλύσουν την κρίση στην Ελλάδα και να αποφύγουν την επιμόλυνση στη ζώνη ευρώ. Όπω και στην Ιρλανδία έχουμε την Τρόικα με του ε, που καθοδηγεί την Ιρλανδική κυβέρνηση και ένας εκπρόσωπος του κόμματος μου στα πλαίσια του σχεδίου αναθεώρησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα βαίνουν αισίως και ότι η Ιρλανδία όντως ε, κάνει πρόοδο, ε, ε, υπάρχει σχετική σταθερότητα και η ανάκαμψη θα είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της γενικότερης οικονομικής ανάκαμψης. Την Τετάρτη αναμένεται στα συμπεράσματα να ανακοινωθεί μια λύση και μια εξαγορά από τον ιδιωτικό τομέα της τάξης του 60%. Εγώ πιστεύω ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει υπό αμφισβήτηση την αγαρογή της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας ε, γιατί δεν μπορεί να επιτρέψουμε 3,4 δις επισφαλών δανείων. Διακόπτεται ο μιλητής από τον Πρόεδρο. Ε, Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Στανόκα τώρα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, 20 χρόνια πέρασαν από τότε που το Ανώτατο Συμβούλιο της Λετωνίας υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο οι πολίτες της Λετωνίας ήταν δεκτοί και μόνο εκείνοι που το 1940 την έδρα τους εκεί και οι απόγονοί τους και βλέπουμε ότι στερήθηκαν πολιτικών δικαιωμάτων Λετών ήταν μοναδική ιστορία στην πρόσφατη ιστορία. Το Κοινοβούλιο αφαίρεσε σημαντικά δικαιώματα ηθαγένειας από τους πολίτες. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Η κατάσταση αυτή όπου οποιοδήποτε υπήκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λετωνία έχει δικαίωμα να ψηφίζει σε ευρωπαϊκές και τοπικές δημοτικές εκλογές. Ταυτόχρονα όμως ένα σημαντικό μέρος των ηθαγενών, των γηγενών και εκείνων που ζούσαν επί δεκαετίες στη Λετωνία δεν έχουν αυτά τα δικαιώματα. Σε σχέση με την πρόταση για την